διανάγνωση για την οδηγία ε, τεχνικέ προδιαγραφέ για τα σκάφη εσωτερική ναυσιπλοεία, τον κανονισμό που αφορά τι κοινοτικέ στατιστικέ για το εξωτερικό εμπόριο, όσον αφορά τι ε, ε, αρμοδιότητε και τι ε, εξουσίε εκτέλεση που έχουν χωριστεί στην Κομισιόν. Οι τίτλοι θα είναι στα πρακτικά. Η τρίμηνη προθεσμία που διαθέτει το Κοινοβούλιο για να εκφραστεί θα αρχίσει να ισχύει από αύριο 23 Ιουνίου.